από την Γκουε Έσοντε ε, ε, Γκουε Άλντε Πράσινους ECR ε, και ΕΛΚ έλαβα τα ονόματα τα οποία προτείνουν για την στελέχωση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπιών. Εάν δεν είχε καμία αντίρρηση, εγκρίνονται. Κυρίες και κύριοι, όπως γνωρίζετε,